οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξ αυτού του θέματος που συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ολοκληρώνεται το θέμα αυτό και θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η σύσταση σε δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα έκθεση του κυρίου Ελκαντράουι. Καταρχάς το λόγο έχει και για τέσσερα λεπτά ο εισηγητής. Ο κ. Σελ Καντράουι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ψηφίσουμε, όπω όπως ελπίζω σύντομα, το κείμενο αυτό που θα είναι μια συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα έχουμε μια σημαντική στιγμή για τον κλάδο των μεταφορών στην Ευρώπη. Ένα πραγματικό ορόσημο για την Ευρώπη η υλοποίηση βεβαίω του οποίου θα εξαρτηθεί και από την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Εμείς εφαρμόζουμε πάντα μία αρχή που για χρόνια υποστηρίζουμε, ότι ο Ριπένων πληρώνει και την αρχή της ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους. Όπως ξέρετε και η προηγούμενη εισηγήτρια κυρία Βότμαν Κόλ είχε αγωνιστεί για το θέμα αυτό το 2008 είχαμε εγκρίνει ένα κείμενο, αλλά έκτοτε καθυστερούσε. Πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ την κατάσταση και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Το τελικό κείμενο είναι συμβιβασμό. Συμβιβασμός και μεταξύ θεσμικών οργάνων και στο εσωτερικό θεσμικών οργάνων. Μικρή είναι η πλειοψηφία που υποστηρίζει το στο κοινοβούλιο τη θέση αυτή. Υπάρχουν αντιστάσεις θεωρούν, κάποιοι θεωρούν ότι είναι πολύ δειλό, άλλοι θεωρούν το κείμενο είναι πολύ φιλόδοξο. Καταφέραμε ωστόσο, πιστεύω εγώ και πιστεύουμε και άλλοι συνάδελφοι, ότι το κείμενο, να φτάσουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο που σας ζητώ να υποστηρίξετε γιατί αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στα κράτη-μέλη πέραν της επιβολής τελών στις υποδομές να λάβουν υπόψη και την ηχορύπανση αλλά και την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται και την δυνατότητα ανανέωσης του στόλου, επιτρέποντας έτσι στα κράτη να εισάγουν μεγαλύτερες μεταβολές, με, με, ε, μεγαλύτερη ποικιλομορφία στην επιβολή τελών χρήσης των οδικών υποδομών. Επίσης οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα τα πράγματα και να αυξήσουν την κινητικότητα. Υπάρχει σαφής δέσμευση, σαφές, σαφέστατη δέσμευση από πλευρά κρατών μελών να επενδύουν εκ νέου τα έσοδα από αυτά τα νέα μέσα σε εξασφάλιση βιώσιμης κινητικότητας και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Επίσης, για το Κοινοβούλιο κάτι πολύ σημαντικό, υπάρχει διαφάνεια ε, στην ε, μορφή αυτή επιβολής τελών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δείξουν ότι χρησιμοποιούν τη διαφάνεια για να υπάρξει ένα αποτελεσματικότερο σύστημα μεταφορών και όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων που καλύπτονται από την οδηγία αυτή να μπορούν να, ε, καλύψουν, να, να, να, να ε, καλύψουν όλους τους μεγάλους οδικούς άξοδους, άξονες. Βασικό χαρακτηριστικό η διαλειτουργικότητα. Χρειάζεται να υπάρχει μία ευρωπαϊκή λύση. Τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω πίνακα αντιστοιχηση. Είχαμε βασικές μεγάλες συζητήσει στο σημείο αυτό. Η λύση που βρήκαμε υπομορφή ε, δηλώσεων των διαφόρων θεσμικών οργάνων είναι νομίζω ικανοποιητικέ. Και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα βρεθεί ευκολότερα λύση. Συνάδελφοι, δεν είναι πανάκια η Ευρωβινιέτα. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της κίνησης. Αποτελεί ωστόσο ένα σημαντικό τμήμα για να φτάσουμε σε ένα σοβαρό, σε ένα πιο ουσιαστικό και ενιαίο σύστημα μεταφορών. Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση βέβαια, χρειάζεται να προχωρήσουμε παραπέρα. Αποτελεί ωστόσο κατά την άποψή μου πρώτο βήμα και γι' αυτό ζητώ να την υποστηρίξετε. Ευχαριστούμε κύριε Ελκαντράουι για το Συμβούλιο το λόγο, έχει η κυρία Γκιόρη. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξέρετε, κύριε βουλευτέ και πρόεδρε, στην αρχή τη Ουγγρική Προεδρία είχαμε υποσχεθεί να εργαστούμε υπέρ μια ισχυρή Ευρώπη. Ευρώπης που στο επίκεντρό τη έχει τον άνθρωπο. Και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να εκδοτήσουμε μία οδηγία χάρη στην οποία θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό χαιρετίζω την συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οδηγία, πάνω στην οδηγία της Ευρωβινιέτας. Αυτή η πρόταση Ε, έχει σαν στόχο τον σωστό καθορισμό των τιμών μεταφοράς, ούτως ώστε το πραγματικό κόστος των βαρέων φορτηγών οχημάτων να υπολογίζεται πλήρως και όσον αφορά τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, πτώσεις της κλιματολογικής αλλαγής κλπ. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι μεταφορές με βαρέα φορτηγά οχήματα είναι απαραίτητη. Από την άλλη μεριά το γεγονός ότι τα προβλήματα που ακολουθούν ε, τις μεταφορές αυτές, δηλαδή ε, συμφόροι στο αυτοκινητόδρομος, ε, ε, της ατμόσφαιρας κλπ. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος διακανονισμός. Μέτρα που έχουν σαν στόχο την εσωτερικοποίηση εξωτερικού κόστου. Ε, πρέπει να είναι όσο πάει και πιο σημαντικά. Δίκες τιμές ε, για τις μεταφορές θα ενθαρρύνουν πιο αηφόρη χρήση των περιορισμένων πόρων. Αυτή η διαχείριση είναι πάρα πολύ σημαντική και υπάρχουν και στη Λευκή Βίβλο που πρόσφατα α, προετοίμασε η Κομισιόν η οποία λέει ότι ένας οδικός χάρτης θα πρέπει να προωθήσει ε, και δίκαιο σύστημα μεταφορών. Αυτό προχωρά προς την επίτευξη του στόχου της εσωτερικοποίησης του πλήρους εξωτερικού κόστους των μεταφορών. Η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα είναι τα πιο σημαντικά στον τομέα των μεταφορών και ξέρουμε ότι ο Κοινοβούλιο συμμερίζει τι απόψει μα. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να πετύχουμε ένα συμβασμό. Η Ουγγρική Προεδρία θα ήθελα να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον εισηγητή τον κύριο Κατραούη για την βούλησή του επικοδομητικής συνεργασίας με το Συμβούλιο. Τα τελικά σημεία των διαπραγματεύσεων ήταν το θέμα των ε, πινάκων αντιστοιχίας. Η Κομισιόν χαιρετίζει το αποτέλεσμα και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μήνυμα της Ουγγρικής Προεδρίας που υποστηρίζουν όμω και οι ρωσικές Προεδρία Πολωνία, ε, Δανία και Κύπρια. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω στα αγγλικά. Δηλώνεται ότι η συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τρεμερή διάλογο 23 Μαου 2011 για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 1999 κάθος 62 ΕΚ για την επιβολή τελών στα βαρέα φορητικά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομή, τη λεγόμενη δηλαδή ευρωβινιέτα, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα των διαθεσμικών συζητήσεων για τους πίνακες αντιστοιχίας. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα έχει σημαντικέ επιπτώσει στην ποιότητα ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ των θεσμικών μα οργάνων και προσβλέπουμε σε μια θετική ψήφο αύριο για το θέμα αυτό που είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ουγγρικής Προεδρίας. Ελπίζουμε ότι τα η πλειοψηφία των μηνών θα υποστηρίξει αυτήν την οδηγία. Σας ευχαριστώ για την φορά για την συνεργασία σας. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τους σκιώδες εισηγητές, τους νομικούς μας εμπεριχνόμενες, ιδίω όσον αφορά το θέμα των πινάκων δυστυχία και του γνώσου πετύχαμε στην συνδεσμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιώργη. Ο Επίτροπος Κάλλης έχει το λόγο. Μετά από διαπραγματεύσεις τριετίες πλησιάζουμε πλέον στην υιοθέτηση της ε, τροποποιωτικής οδηγίας, της λεγόμενης οδηγίας ε, Eurovignette. Είναι τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής για εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών σε όλα τα είδη μεταφορών. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βελγική Προεδρία που ξεμπλόκαρε το θέμα στο Συμβούλιο. Η Ουγγρική Προεδρία με μεγάλη ικανότητα διαπραγματεύτηκε και πέτυχε την απαιτούμενη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερα τον εισηγητή κύριο Ελχαντράουι, ο οποίος μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βελτίωσε το κείμενο στη δεύτερη ανάγνωση. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει την οδηγία αυτή για δύο λόγους. Πρώτον, για να πετύχουμε του στόχου μα για ένα πράσινο σύστημα μεταφορών, περισσότερο αηφόρο, και να εφαρμόσουμε την αρχή του όποιος μολύνει πληρώνει. Η οδηγία θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν τέλη στα φορτηγά όχι μόνο για το κόστος των υποδομών που χρησιμοποιούν όπως ισχύει σήμερα, αλλά και για τον θόρυβο και τη μόλυνση του ε, αέρα. Αυτό θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες ώρες. Δεύτερον, σε, μια εποχή όπου δεν υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα, η οδηγία αυτή θα δημιουργήσει νέα έσοδα και θα καταστήσει νέους πόρους διαθέσιμους για υποδομές στον τομέα των μεταφορών. Υποστηρίζει η Επιτροπή τη συμφωνία αυτή. Άκουσα αυτά τα οποία είπατε για τους πίνακες αντιστοίχησης. Ελπίζω να συμφωνήσουμε. Ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να κάνω την επίσημη δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει την ανηλυμένη της υποχρέωση για την δημιουργία πινάκων αντιστοίχησης σχετικά με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια της μεταφοράς της κοινοτικής οδηγίας στις διάφορες χώρες προς όφελος των πολιτών, προς όφελος της διαφάνειας και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην εξέταση της συμβατότητας των εθνικών ρυθμίσεων με τις ευρωπαϊκές προβλέψεις. Λυπάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έλλειψη υποστήριξης κάποιων προτάσεων από πλευράς ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την 1099 ε, κάθετος 62 για τη χρήση ορισμένων υποδομών. Κάτι το οποίο θα καταστήσει, θα έλεγα, την χρήση των πινάκων αντιστοίχησης πλέον υποχρεωτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια ενός πνεύματο συνεργασίας και για να διασφαλίσει την άμεση υιοθέτηση αυτής της πρότασης δέχεται την αντικατάσταση των υποχρεωτικών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στου πίνακε με το νέο κείμενο και ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πρακτική. Θα ενημερώσει 12 μήνε μετά την υιοθέτηση τη συμφωνία αυτή στην Ολομέλεια για την εξέταση των πραγμάτων και θα κάνει και μια έκθεση στο τέλος της μεταβατικής περίοδου της πρακτικής αυτής των κρατών μελών έτσι ώστε ελπίζουμε οι πίνακες αντιστοίχησης να δείχνουν ακριβώς τις αντιστοιχίες που υπάρχουν ανάμεσα στα εθνικά μέτρα και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο συγκεκριμένο θέμα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν προηγούμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της έτσι ώστε να βρει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια κατάλληλη λύση σε αυτό το οριζόντιο θεσμικό πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στις πολιτικές ομάδες. Για το ΕΛΚ και για δύο λεπτά η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η οδηγία για την Ευρωβινιέτα είναι σημαντική γιατί θέτει ευρωπαϊκούς κανόνες παιχνιδιού για τον καθορισμό του κόστους ένα χιλιόμετρο. Άρα περιορίζει το περιθώριο δράσεις ε, στο εσωτερικό της Ένωσης δίνοντας ακριβώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Και η πρόταση της Επιτροπής και η θέση του εισηγητού σε πρώτη ανάγνωση ε, δεν ήταν επαρκώς φιλόδοξη. Ωστόσο, ε, ο εισηγητής, ευτυχώς ο εισηγητής, πέτυχε σημαντική πρόοδο φτάνοντας κοντά στις θέσεις μας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ ιδίω στη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου, παρά, που παρά την εσωτερική σύγκρουση στο Συμβούλιο, κατόρθωσε να πετύχει μια στέρεη πλειοψηφία και κάτι που αντικατοπτρίζεται και στη στέρεη πλειοψηφία και στο Κοινοβούλιο. Εμείς θα υποστηρίξουμε το συμβιβαστικό κείμενο που δίνει τα πρώτα βήματα για την ε, οριστική υλοποίηση της αρχής του οριπένων πληρώνει. Κάτι πολύ λογικό άλλωστε ενισχύονται ταυτόχρονα, προστίθενται κίνητρα για τη βιωσιμότητα. Επιβάλλονται ε, ε, ε, σημαντικότερα τέλη σε ώρες εχμής για καλύτερη διαχείριση των συνθήκων κυκλοφορίας. Ορίζονται καλύτερα οι ώρες εχμής. Είναι θεμελιώδες επίσης το αίτημα της αντιμετώπιση ολόκληρη τη διαλογικότητα του συστήματο, κάτι που δεν είναι ακόμα ε, εξασφαλισμένο. Επίση, το ER marking είναι σημαντικό, δηλαδή ο συγκεκριμένο στόχο των πόρων για το Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό επίση, είναι η ανάγκη των υποχρέωσεων των κρατών να αναφέρουν που χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι αυτοί. Για δύο λεπτά για τους σοσιαλιστές και δημοκρατές ο κύριος Ερτούγκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Μετά από ένα μακρύ μαραθώνιο διαπραγματεύσεων κατάφερε ο συνάδελφος Ελκατροή και εκπρόσωπο του Συμβουλίου και της Κομισιόν να ε, κρίνουν ένα πακέτο για τη χρήση βαρέων φορτηγών οχημάτων στην Ευρώπη. Για όλα αυτά είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον εισηγητή μας. Η αρχή της εσωτερικοποίησης των εξωτερικού κόστους με εν μέρη δέσμευση των πόρων που εισπράττονται για την προώθηση των δεδομένων και την χορήγηση κινήτρων είναι σημαντική στόχη για την επίτευξη του Λευκής Βίβλου Μεταφορών. Επίσης νομίζω ότι το θέμα της διαφάνειας είναι κάτι που πρέπει να ισχύει και να επιβάλλεται και από το Συμβούλιο τα κράτη-μέλη ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της, ε, ε, των διαπραγματεύσεων <clears throat> τριμερούς διαλόγου προσπάθησαν λέω να μπλοκάρουν ε, την οδηγία μέσω των πινάκων αντιστοιχία. Αυτό δεν είναι κακό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους να δεχθούν τον ευρεθέντα συμβασμό και να μην διακυμεύσουν τις διαπραγματεύσεις. Γιατί αυτό θα βοηθήσει εκείνους που δεν θέλουν να προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ελτούκ. Για δύο λεπτά για τους φιλελεύθερους και δημοκράτες ο κύριος Στέρξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Παρά την σημαντική προσπάθεια του εισηγητού που συγχαίρω γι' αυτό, το κείμενο πόρο απέχει από το να είναι τέλειο. Ιδίω για την δεσμευτική χρήση των πόρων. Τι νόημα έχουν τα τέλη να κάνουν βιώσιμες και ορθολογικές τις οδικές μεταφορές. Αυτό δεν το επιτυχάνουμε απόλυτα. Επίσης, τα κράτη-μέλη κρατούν τη δυνατότητα να μην περιορίζουν το εξωτερικό κόστος. Η, εσωτερική, η ενσωμάτωση λοιπόν δεν σημαίνει πλήρη κατάργηση. Τα κόστη αυτά μπορούν να παραμείνουν έξω. Επίσης, λείπει κάτι κατά την άποψή μου. Αν επιβάλλουμε διαβάθμιση των τελών για τις ώρες εχμής, πλήττουμε τα θύματα των ουρών, όχι αυτούς που δημιούργησαν τις ουρές. Στην πρώτη ανάγνωση υπήρχε ένας ειδικό πίνακας, ο οποίος καθοδόν χάθηκε. Ο εισηγητής θα πρέπει να εξηγήσει κατόπιν πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων που εισπράττονται με τον τρόπο αυτό. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ του κλάδου και των αρμόδιων αρχών για να υπάρξει ένας ορισμός του τι είναι στοχοθετημένες επενδύσεις. Η έκθεση, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικ... έχει σημαντικά κενά, αλλά αποτελεί πρώτο βήμα. Μπαίνουμε σε έναν πρώτο υπολογισμό του εξωτερικού κόστους και μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε την βιωσιμότητα και την ε, ε, ευκολία κυκλοφορία. Η Λευκή Βίβλο υπογράμμιζε την ανάγκη κάτι τέτοιο. Αν δεν δεχθούμε λοιπόν την έκθεση αυτή, θα μπλοκάρουμε και μια σειρά άλλων βημάτων και θέσεων που προτείνει η Λευκή Βίβλο. Για το λόγο αυτό ήταν δύσκολο να υπάρξει συμφωνία για το ζήτημα. Όπως ανέφερα, αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα. Ευχαριστώ για τους συντηρητικούς ο κύριος Ζήλε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Προεδρία και τον Επίτροπο. Κυρίες όμως φυσικά να ευχαριστήσω τον κύριο Αλκαντράουι για μια πολύ κανή διαπραγματευτική τακτική που ακολούθησε. Πολλές από τις λύσεις στις οποίες καταλήξαμε είναι πάρα πολύ καλές. Να ενθυμούμεθα ότι ο συμβιβασμός στο Συμβούλιο ήταν πάρα πολύ εύθραστος και το θέμα της εμβέλειας της οδηγίας, όπως επίσης και της χρήσης των προσόδων, ήταν κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα αμφισβητήσιμο. Και πολλοί πιστεύαμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγούσαν σε χειρότερες λύσεις και σε καθόλου λύσεις. Η εφαρμογή του όποιος ρηπαίνει πληρώνει της αρχής αυτής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι δεδομένο πλέον. Η βασική αυτή αρχή, όπως επίσης και τα τέλη, θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες μέλη. Δυστυχώς πάρα πολλές δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα τις υποδομές γύρω, το θέμα μάλλον των τελών, το λεγόμενο Eurovinet 1. Είναι πάρα πολύ πίσω και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα ανταγωνισμού. Αν γίνουν σεβαστοί οι κανόνες, χρησιμοποιώντας με σωστό τρόπο τα χρήματα του φορολογούμενου, τότε ε, το εξωτερικό κόστος δεν αντισταθμίζεται. Ευχαριστώ κύριε Τσίλε. Για τους πρασίνους τώρα, κυρία Λίχτενμπεργκερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Συνάδελφοι, η Ευρωβινιέτα είναι παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το, το Συμβούλιο προσπαθεί να μπλοκάρει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου σε μια σειρά θεμάτων. Έχουμε μια πολιτική μεταφορών που πρέπει να μας έπε, που έπρεπε να μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όμως κάτι σαφές είναι ότι υπάρχει κόστος για την ρήπανση πέραν της ηχορήπανσης και το κόστος το πληρώνει όχι ο ρηπαίνων αλλά ο καταναλωτής. Καταφέραμε τελικά να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των διαφόρων χωρών. Το κείμενο αυτό αποδυναμώθηκε ωστόσο περαιτέρω Φερρυπίνη. Ο υπολογισμό του εξωτερικού κόστου γίνεται σε θελούσια βάση. Το κόστο δεν καλύπτει όλες τις ε, μορφές ρήπανσης, κάποιες μόνο, ενώ επιπλέον το μένουν πολύ λίγα πράγματα. Πέρασε η Γερμανία τη θέση της για τους 12 τόνους, ενώ για τις ορεινές περιοχές δεν καλύπτουμε τα μεγαλύτερα φορτηγά. Η Ιταλία έχει μια σειρά προβλημάτων που δεν τα άφησε να περάσουν και αυτός είναι ένας τρόπος που δείχνει ότι δεν λαμβάνουμε παρκώς υπόψη όλες τις διαστάσεις των μεταφορών. Πάντως, η βασική αρχή της, του υπολογισμού των του εξωτερικού κόστους λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ. Για τους για 1,5 λεπτό για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά ο κύριος Κόλιτσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Η οδηγία Eurovignette είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε λήψη μέτρων διακόπτειο. μιλητής. Λοιπόν, επαναλαμβάνει ο, ομιλητής, Η οδηγία Eurovignette, λοιπόν είναι τμήμα των οδηγιών που θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εξομάλυνση των συνθήκων μεταφορών. για τις ιοδρομικές μεταφορές οι πληρωμές από πλευρά του κοινού είναι δεδομένες, αλλά για τις οδικές μεταφορές οι πληρωμές είναι σε συμβολικό επίπεδο στις περισσότερες χώρες. Ιδιαίτερα στα βαρέα οχήματα βλέπουμε ότι οι υποδομές οι οποίες είναι οι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του τύπου αυτού των μεταφορών είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οπότε πάρα πολύ σωστά Κατά συνέπεια μάλλον οι τοπικές αρχές εκεί όπου υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι υφίστανται την μεγαλύτερη βλάβη. Εδώ εφαρμόζεται πάντως για πρώτη φορά με συνολικό τρόπο η αρχή του όποιος ρηπαίνει πληρώνει. Έτσι προσπαθούμε να εσωτερικεύσουμε το εξωτερικό κόστος των μεταφορικών δραστηριοτήτων. Είμαι πάρα πολύ περίεργος για να δω πώς τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 που δεν είναι παρά ένα χλωμός καθρέφτης του τι χρειάζεται πράγματι η ε, δραστηριότητα αυτή. Υποστηρίζουμε πάντως τη θέση του κυρίου Ελχαντράουι. Ευχαριστούμε κύριε Κόλιτσεκ. Κάποιος σήκωσε μπλε κάρτα. Κύριε Λάιτφριτ, συμφωνείτε. Señor ε, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Κύριε Κόλισε. συμφωνείτε να ακούσετε την ε, παρατήρηση με τη διαδικασία της μπλε κάρτας από τον κύριο Λάιξφελτ. Έχετε το λόγο. Κύριο κύριος ε, Κόλιτσεκ, δεν ξέρω, μήπως δεν σας κατάλαβα καλά, αλλά ήθελα λιγάκι να διευκρινιστεί το θέμα. Νομίζω ότι είναι σχετικά σαφές ότι αυτή η συμβαστική πρόταση είναι αδύναμη και η πρόταση σχετικά με τα φορτηγά στους δρόμους εξακολουθεί να υφίσταται και τα διόδια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Εσείς είπατε ότι με αυτήν την οδηγία επιτυγχάνεται κάποια ισορροπία ανάμεσα στις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Εγώ δεν είμαι ευτυχισμένο γι' αυτό, αλλά ενδέχεται να μην σα κατάλαβα καλά. Έχετε την καλοσύνη παρακαλώ να διευκρινίσετε. Ο κύριος Κόλιτσεκ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για εξομοίωση κατά κάποιο τρόπο των διαφόρων συνθήκων. Γιατί στις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές εμ, επιβάλλονται τέλη για τη χρήση των υποδομών. Και επαναλαμβάνω και στα γερμανικά, αυτό είναι το πρώτο βήμα για εξομοίωση των όρων μεταξύ σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Γιατί μέχρι στιγμή. Καταβάλλονται τέλη για τι σιδηροδρομικέ υποδομέ, αλλά ελάχιστα καταβάλλονται για τη χρήση των οδικών υποδομών. Είναι το πρώτο βήμα, ένα ελάχιστο βήμα για την εξομοίωση των συνθηκών μεταξύ οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, επαναλαμβάνω. Εκ μέρου ε, τη ε, Ευρώπη ε, Δημοκρατία και Ελευθερία, ο κύριο Ιμπράστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το αξιόλογο έργο που επιτέλεσε. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο και στην κινητικότητα και στην ε, οικονομική ανάπτυξη και θέλουμε να ευνοήσουμε το, την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα θα πρέπει να αποσυμφορήσουμε τις οδικές μεταφορές. Να έχουμε επίγνωση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν και εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Υπάρχουν και περιβαλλοντικέ συνέπειε και συνέπειε στη δημόσια υγεία και όλα αυτά συνδέονται με την ορθολογική χρήση των μεταφορών. Και η εφαρμογή τη αρχή ορυπαίνων πληρώνει θα πρέπει να μα οδηγήσει στη λήψη μέτρων προκειμένου να περιορίσουμε τη ρήπαση του περιβάλλοντος, την ηχορύπανση, την σπήλωση του τοπίου και τις αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Βέβαια, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναλάβουμε το σημαντικό οικονομικό κόστος όλων αυτών των μέτρων και θα πρέπει να το επιρρύψουμε στους ε, ώμους των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι σημαντικό να είμαστε αποφασισμένοι και να εφαρμόσουμε αυστηρά την αρχή ορυπαίνων πληρώνει και δεν αφιβάλλω ότι αυτό θα μεταφραστεί σε θέσπιση πιο αποτελεσματικών μέτρων ε, επιβολής τελών στις μεταφορές ή θα δημιουργηθούν ε, πιο αποτελεσματικά συστήματα προσφοράς και ζήτησης. Τα σημερινά όμως μέτρα δεν είναι τα πλέον κατάλληλα και θα ευνοήσουν μόνο ορισμένα κεντρικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ε, χώρες διαμετακόμισης. Τέτοιου είδους μέτρα όμως δεν ευνοούν καθόλου πιο περιφερειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτό το στοιχείο και να τα εξετάσουμε υπό διαφορετικές σκοπιές πριν εγκρίνουμε τελικά αυτά τα μέτρα. Εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων για 1,5 λεπτό κύριο Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, λέει, να αυξήσει τα έσοδά της φορολογώντας τα φορτηγά. Ωραία. Θα ρωτήσω και όταν ρωτώ μάλλον τους εκλογείς μου τι πιστεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μου απαντούν ας μην μπούμε καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός ε, ε, από ε, τα προβλήματα που είχαμε με την κατασκευή φορτηγών μέχρι να φτάσουν σε εμά, τώρα έχουμε και τη φερολογία. Η τηλεόρασή μας δεν δείχνει την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνο σαπουνόπερες. Δεν πουλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν είναι είδηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα φορολογούμε λέει και τα φορτηγά για τα διευρωπαϊκά δίκτυα λέει των μεταφορών ε, που συμπεριλαμβάνουν και τρένα υψηλής ταχύτητας. Δηλαδή, όταν αυξάνονται οι φόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι γίνεται, τίποτα, γιατί ο κόσμος δεν έχει ιδέα. Το υπερκράτος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, κάνει τους πολίτες άβουλους υπνοβάτες, αδιαφορεί ο τύπος και το Ηνωμένο Βασίλειο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Σας ευχαριστώ κύριε Νάτρας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι ομιλητές τώρα. Για δύο λεπτά ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να συγχαρώ και τους συναδέλφους για τη δουλειά τους. Γιατί δεν ήταν εύκολο να αναζητηθεί ο συμβιβασμός. Πολλοί ε, που βρίσκονται εδώ βεβαίως δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Θα ήθελα όμως ευθύς εξ αρχής ε, να πω προειδοποιητικά το εξής. Αυτοί που περιμένουν περισσότερα, αν αυτοί ε, κάνουν συμμαχία με αυτούς που περιμένουν λιγότερα και τελικά αποτύχει το όλο εγχείρημα, θα είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω όσοι επιθυμούν την συμπερίληψη του κόστου να στηρίξουν αυτό το συμβιβασμό. Σε μεγάλο βαθμό αυτή είναι η θέση του ΕΛΚ, αν και δεν συμφωνούν με αυτή όλε τι αντιπροσωπείε ε, που ε, βρίσκονται στο ΕΛΚ. Εμεί ε, είμαστε υπέρ του να χρησιμοποιήσει κανείς μέσα για την κινητικότητα. Και αυτό για μας είναι από τα σημαντικότερα σημεία. Όπως αναφέρθηκε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να καταστήσουμε ακριβότερες τις μεταφορές, γιατί αυτό δεν είναι αποδοτικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ισορροπία και ε, να μπορούν να γίνουν επενδύσεις στα μέσα της ε, κινητικότητας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για μας είναι η διαλειτουργικότητα. Τα συστήματα της ε, χρέωσης χρήσης δρόμων, τα διόδια δηλαδή, Δηλαδή ε, δεν θέλουμε να τα θέσουμε σε κίνδυνο επειδή υπάρχουν 27 διαφορετικά συστήματα. Ε, κατόπιν τούτου το Συμβούλιο πρέπει να είναι λιγάκι περισσότερο ευέλικτο από ό,τι ήταν κατά παρελθόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι να υπάρχουν φορτηγά φιλικά προς το περιβάλλον. Άρα δηλαδή και εδώ πρέπει να καταδείξουμε τη σωστή κατεύθυνση και αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως όλα όσα προβλέπονται δεν είναι υποχρεωτικά. Άρα όσοι ε, είναι υπέρ της συμπερίληψη του κόστου, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί και εγώ προσωπικά θα επιθυμούσα όλα αυτά να γίνουν δεσμευτικά στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτή η συζήτηση έχει γίνει επανειλημμένα στο Κοινοβουλίο. Τι θέλουμε, 27 διαφορετικά διόδια ή θέλουμε όλα τα κράτη να έχουν ένα ενοποιημένο σύστημα. Και μήπω θεωρείτε ότι πρέπει να προκύψει κρίση για να αρχίσουν πάλι όλοι να κάνουν έκκληση στην Ευρώπη. Μα μόνο η Ευρώπη θα φέρει τη λύση και όχι τα διαφορετικά συστήματα διοδίων στις διάφορες χώρες. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Το λόγο έχει ο κύριος Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε. Κοιτάξτε, στη συζήτηση αυτή υπάρχει ε, κάποιος ε, που ε, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αυτός είναι ο εισηγητής. Πραγματικά εγώ πιστεύω ότι ο εισηγητής σε, αυτό το θέμα ε, μπόρεσε να ξεπεράσει πολλά ανυπέρβλητα εμπόδια και κατόρθωσε να επιτύχει το μέγιστο. Πράγματι, εδώ στο Κοινοβούλιο δεν υπάρχει πλειοψηφία για μια ε, πραγματική οικολογική διαμόρφωση των μεταφορών. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και είναι απόλυτα σαφές ότι αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο υπάρχει μια πλειοψηφία Υπουργών Μεταφορών που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το περιβάλλον. Υπάρχει μια πλειοψηφία στο Συμβούλιο που αδιαφορούν παντελώς ε, για όσους ε, βρίσκονται πάνω σε δρόμους μεταφοράς. Ε, οι υπουργοί τελικά δεν ενδιαφέρονται στο να αγοράζουν οι καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα αν λάβει κανείς όλα αυτά υπόψη του, νομίζω ότι επιτεύχθηκε το μέγιστο. Γιατί υπάρχει καταρχήν η αρχή του εξωτερικού κόστους. Αυτό είναι ένα δύσκολο βήμα, αν λάβει κανείς υπόψη του την αντίδραση. Για πρώτη φορά λοιπόν ε, μας προσφέρει τη δυνατότητα ε, τις εκπομπές να τις ε, χρεώνουμε. Βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ λίγα, αν δει κανείς την κατάσταση. Ίσως πράγματι να πρόκειται για σταγόνα εν το ωκεανό. αυτό το οποίο επιτεύχθηκε είναι και να διευρυνθούν οι διάδρομοι. Όμω δεν κατέστη δυνατόν να χρεώσουμε πραγματικά, ουσιαστικά τι εκπομπέ διοδίων. Μα οι οδικέ μεταφορέ είναι από, τους, από τις μεγαλύτερες πηγές ρήπανση στην Ευρώπη και δεν χρεώνονται. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ με του συναδέλφου εκείνου που λένε ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε γιατί αλλιώ θα καταστραφούν τα πάντα. Βαριά την καρδία το πράτο αυτό ε, και θεωρώ καλά κάναμε που φτάσαμε μέχρι εδώ, όμω θεωρώ ότι στο μέλλον πρέπει να βελτιωθεί πολύ περισσότερο η κατάσταση. Για 1,5 λεπτό το λόγο κυρία Μάισνερ. Κυρίες και κύριοι, ο Επίτροπος κύριος Κάλλας στη Λευκή Βίβλο περιγράφει διάφορα πράγματα για τα πώς οραματίζεται το μέλλον. Λέει ότι χρειάζονται κίνητρα για να υπάρχουν μεταφορές φιλικότερες προς το περιβάλλον και λέει επίσης ότι χρειάζονται και νέες πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε να ισχύει η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Η αεροβινιέτα που, για την οποία μιλάμε σήμερα είναι ο δρόμος εκείνος που μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε και τα δύο και πρέπει να πω ότι ε, αυτά όλα ξεκίνησαν με τη Βελγική Προεδρία. Ε, τότε είχαμε τρεις ε, σημαντικές ε, προσωπικότητε εκτός Βελγίου και τον εισηγητή τώρα που κατόρθωσαν πραγματικά να ανοίξουν ένα νέο δρόμο για να ζητηθούν νέοι δρόμοι. Βεβαίω θέλω να πω ότι εγώ θα επιθυμούσα αυτή η βελγική πράξη να στεφτεί με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι υπάρχει σήμερα γιατί είναι ένα μικρό συμβασμό αυτό που πετύχαμε. Εν πάση περιπτώσει τώρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο στόχο το 15% του κόστου των υποδομών και το 15% ε, του ε, εξωτερικού κόστους ε, θα πρέπει να συνυπολογίζεται. Ίσως να είναι λίγο αυτό. Όλοι οι πολιτικοί των κρατών μελών λένε ότι χρειαζόμαστε μέσα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα δίκτυα υποδομών και βεβαίω τα κονδύλια θα πρέπει να πλέξουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, όμως η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που μπορεί να βελτιωθεί υπεραιτέρω στο μέλλον και γι' αυτό το λόγο όλοι λέμε ότι επιθυμούμε να στηρίξουμε αυτή τη συμβαστική πρόταση. Σκληρή η διελκυστίνδα, ίσω να μην είχαμε πετύχει και τίποτα, γιατί ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούν να μην υπάρξει τίποτα. Κατόπιν τούτου, αυτό που έχουμε σήμερα θεωρούμε ότι είναι επιτυχία και θα το υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Το λόγο έχει ο κύριος Βλάσακ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η οδηγία αυτή, την οποία Παρουσίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σχεδιάζει ε, την επιβολή ε, διοδίων σε κάποια φορτηγά βάσει της αρχής ορυπαίνουν πληρώνει γιατί πληρώνουν με πολλαπλούς τρόπους και με ηχορύπανση και με την εκπομπή των καυσαερίων και αυτό έχει επιπτώσεις και στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη χρησιμοποίηση όλων των μέσων μεταφοράς. Ε, και σε τοπικό επίπεδο. Ας πούμε, στις πόλεις είναι πολύ αρνητικές επιπτώσεις και επειδή έχουμε τώρα και την οικονομική κρίση και ε, επιβάρυνση επιπλέον των ε, μεταφορέων, είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να υπάρχει μία περίοδος σταδιακής επιβολής αυτού του τέλους ανανέωση του στόλου ας πούμε. Θα πρέπει να δίνονται κίνητρα για επενδύσεις σε πιο οικολογικά αυτοκίνητα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Τζιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μα σήμερα δεν χρειάζεται να χαιρόμαστε. Απέχουμε πόρο από μια οικολογική ε, κατάσταση στις μεταφορές, ένα σύστημα όπως είπαν κάποιοι. Το κείμενο αυτό τι επιτρέπει. Επιτρέπει απλώς ε, τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα εθελοντικά να χρησιμοποιούν το σύστημα ρηπαίνων πληρώνει. Δίνει την άδεια στα κράτη-μέλη να το ε, πράττουν αυτό. Αλλά είναι τέτοιο στενός κορσές που τελικά ε, θα στοιχήσει άντε τρία ή τέσσερα σέντς παραπάνω. Ε, και αυτό πώς θα είναι κίνητρο για να αλλάξουμε τρόπους μεταφοράς. Δεν είναι καθόλου επιτυχία οικολογική αυτή. Αυτή ήταν η περίφημη εσωτερήκευση ε, του κόστους ε, παρόλα τα όσα έπραξε και ο εισηγητής και το Συμβούλιο. όλα αυτά, επαναλαμβάνω, εμείς θα υπερψηφίσουμε την αρχή αυτή γιατί είναι σημαντική, το είπαν και άλλοι, όπως και την αρχή της προφύλαξης που στις ευρωπαϊκές οδηγίες επέτυχε, αλλά τώρα συζητάμε μόνο για μία αρχή. Παραμένει η μάχη ακέραια, θα πρέπει να τη δώσουμε για να έχουμε πιο οικολογικές μεταφορές, καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Στάσεν. Πρόεδρε, η σημερινή πρόταση για την Ευρωβινιέτα Ε, σε τι καταλήγει η ε, αποτελεσματική τρόποι μεταφοράς που είναι οδική μεταφορά θα χρηματοδοτήσουν τον αναποτελεσματικό σιδηρόδρομο. Είναι ένα βήμα, αλλά βήμα στη λάθος κατεύθυνση. Εθελοντική σήμερα η συμμετοχή ε, των κρατών, αλλά σε λίγο θα γίνει υποχρεωτική. Και σήμερα την πληρώνει το φορτηγό, αύριο θα την πληρώσει το γιοταχή. Οι μεταφορικές ε, ε, εταιρείε. Καλό είναι να ετοιμαστούν να βάλουν στα φορτηγά του εκεί στην καμπίνα του οδηγού και ένα ταμείο τώρα για να πληρώνουν μια στιγμή διακόπτει ο πρόεδρος. Κυρία Στάσεν, σας παρακαλώ, θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά, διότι δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς μα. Λίγο πιο αργά, για να σας καταλάβουμε. Μάλιστα. Πρόεδρε, έλεγα λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πρόταση αυτή ε, θέλει να καταπνίξει και να σκοτώσει ουσιαστικά το κλάδο των οδικών μεταφορών με πρόσχημα την κλιματική αλλαγή. Και μάλιστα τελικά όλα αυτά θα είναι αναγκαστικά για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στάσεν. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Καντσάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Ε, πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω την εργασία του εισηγητή κυρίου Καντράου και τον συγχαίρω γι' αυτό γιατί ε, πραγματικά ε, προσπάθησε να βρει κάποιο συμβασμό προσπάθησε σκληρά και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη στην τελική συμφωνία μάλλον θεωρώ ότι το θέμα αυτό θα πρέπει ε, να ακολουθεί ε, τον δρόμο της ε, συνδιαλλαγής. Δυστυχώς εδώ δεν πρόκειται για λεπτομέρειες όπως αναφέρθηκε. Η αρχή ότι ο ρηπαίνων πληρώνει είναι σωστή αυτή η αρχή και τη συμμεριζόμαστε και μόνο για να καταστούν οι μεταφορές φιλικότερες προς το περιβάλλον υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Αυτό όμως το εργαλείο που επιλέγεται, η είναι μεροληπτικό αυτό το μέτρο και α μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Κατόπιν τούτου το να θίξουμε μια οικονομική κατηγορία πολύ σημαντική για την αγορά μα, αυτό είναι λάθο. Ε, καλύτερα να δούμε πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα έστω και σε κάποιο μικρό βαθμό για τις υποδομές. Εγώ ε, θεωρώ ότι υπάρχει ένας πολύ περίπλοκος μηχανισμός υπολογισμού γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι επικριτικός απέναντι σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι η πρόταση τιμωρεί ε, απαράδεκτα ε, τις χώρες εκείνες ε, που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού δεν είναι δεδομένη και αυτή η ροή των μεταφορών δημιουργεί ε, προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα τώρα και άλλα που θα προκύψουν στο μέλλον εάν συνεχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο χρέωσης. Εγώ θεωρώ ότι τα κράτη είναι ελεύθερα να χρησιμοποιούν το σύστημα της προσάυξησης. Όμως όσον αφορά ε, το θέμα των μεταφορών εξαρτώμεθα όλοι μεταξύ μας ο ένας από τον άλλο. Η επιτυχία με κάθε τίμημα αυτή αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν, κυρίως όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής αυτών των προτάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά το λόγο η κυρία Γιάλα. Γιάλα. Η ε, κυρία Γιάλα. Συγγνώμη. Μόλις με είχα φωνάξει και ήμουν έξω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την αποφασιστικότητα και την πυγμή του εισηγητή Ελχαντράουι. Πάντως ήθελα να πω ότι οι ιδιαίτερες περιστάσεις των περιφερειακών χωρών που δεν έχουν εναλλακτική λύση για τις, από τις οδικές μεταφορές ε, δημιουργεί προσκόμματα. Για παράδειγμα έχουμε στα, στα Πυρηναία πολλά προβλήματα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας για να έχουμε βιώσιμες σιδηροδρομικές μεταφορές εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ο κύριος Κάλλας ότι ε, αφιβάλλει για την πιθανότητα διάβασης μέσω των ε, πυρηναίων ε, για την επόμενη περίοδο. Οπότε δεν υπάρχει εναλλακτική ως προς τις οδικές μεταφορές και με την Ευρωβινιέτα επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο τις οδικές μεταφορές που είναι οι μοναδικές που χρησιμοποιούν οι περιφερειακές χώρες για τη μεταφορά τροφίμων. Άλλωστε είναι δύσκολο να μεταφέρουμε στους μεταφορείς μια τέτοια δυσάρεστη είδηση ε, επιβάρησης. Βέβαια η κυρία Τυρών είπε ότι τέσσερα ε, εκατοστά δεν είναι τίποτα, αλλά μετά την κρίση που είχαμε με τα αγουράκια και μετά τις ανεύθυνες ε, και χωρίς αποδείξεις, κατηγορίες που έπληξαν βάναυσα την Ισπανική Γεωργία, αλλά όχι μόνο τη Γεωργία και της μεταφοράς. Αυτά λοιπόν τα λίγα δέκατα του ευρώ θα δημιουργήσουν μεγάλες μεγάλα προβλήματα και επιβάρηση στους ε, Ισπανούς μεταφορές, στους Ισπανούς μεταφορείς. Παρ' όλα αυτά θα ήμασταν διατεθειμένοι, ε, κύριε Χαδράου, από την αρχή, από την αρχή που έγιναν οι πρώτοι λογαριασμοί και είδαμε ότι με την επιβάρηση αυτή, με τα τέλη, αυτή, αυτά θα είχαμε προβλήματα, ε, είχαμε αφαίρεση ορισμένων στοιχείων. Γιατί αφαιρέθηκαν. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά πάντως, παρά τα προβλήματα που επισήμανα, θα ήμουν έτοιμη να κάνω κάποιες θυσίες αν επιληθούν σημαντικά προβλήματα, όπως η συμφόρηση. Αυτή τη στιγμή όμως η συμφόρηση δεν περιλαμβάνεται. Άλλο σημαντικό πρόβλημα, η κατάσταση των αποδομών και η ανάγκη βελτίωσης των αποδομών για να βελτιωθεί και η χορύπανση, να περιοριστεί η χορύπανση. Αλλά ούτε γι' αυτό υπάρχει αναλεκτική λύση, δεν υπάρχουν ε, μέτρα κατάλληλα για την καταπολέμηση της. Γι' αυτό η, σοσιαλιστική, η, ισπανική αντιπροσωπεία των σοσιαλιστών είναι υποχρεωμένη να καταψηφίσει την έκθεση. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο κυρία Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ. Δύο λόγια μόνο για να συνοψίσω το γενικό ύφο που επικρατεί στη συζήτηση. Δεν ήθελα να πω ότι τελικά και κρίμα μετά από χρονοβόρε διαπραγματεύσει καταλήγουμε σε συμβαστική λύση και η αρχή ορυπαίνων πληρώνει, αρχίζει και λαμβάνει σάρκα και οστά και στην περίπτωση αυτή. Είναι όμω κρίμα γιατί παρόλο που είναι περίπλοκα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά πολλών χωρών μελών, θα έπρεπε πάση θυσία να είχαμε προσπαθήσει να αφιερώσουμε τα έσοδα στις επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Κύριε Κάλλας, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει αυστηρό έλεγχο. Κρίμα, γιατί καταλήξαμε στη συμφωνία ελαχίστων σε ό,τι αφορά την επιθυμία αποσυμφόρησης. Γιατί ναι, μεν ε, κρατάμε την ε, έννοια των ορών ε, που δεν επίπτουν σε ώρες αιχμή, παρόλα αυτά είναι αρκετά χαλαρές οι διατάξει που προτείνουμε. Και εκεί θα πρέπει την όθηση να τη δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τρίτον, παρόλο που η οδηγία μιλάει για τα βαρέα οχήματα 3,5 τόνων από το 2012 και συμπερίληψη του στη συμφωνία, η δυνατότητα εξαίρεσης είναι μια πολύ επιζήμια υποχώρηση που κάνουμε και θα πρέπει και πάλι εκεί να πρωτοστατήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μικρός συμβασμός, τριοπαθές και καθόλου φιλόδοξο το βήμα, αλλά είναι παρόλα αυτά ένα βήμα και θα το υπερψηφίσουμε. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τσαρνέτσκι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ είπε ότι είναι πολύ ορθολογικές αυτές οι διατάξεις ε, και θα πρέπει να ε, δώσετε ονόματα για αυτούς που πιστεύουν ότι οικονομικά δεν θα έχει προβλήματα αυτή, ε, αντίκτυπο αυτή η διάταξη. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές επίμαχες διατάξεις σε αυτήν την πρόταση. Γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα στις ε, εταιρείες μεταφορών βα, βαρέων οχημάτων. Και πού θα πάνε όλα αυτά τα, χρήματα που θα συλλέξουμε από τα τέλεια, σε ανόητα σχέδια κάποιων περιθωριακών ομάδων. Θα πρέπει να επαναχρηματοδοτηθούν στις οδικές μεταφορές, στη βελτίωση των αποδομών. Αυτό θα το καταλάβαινα. Να γίνει πραγματική αξιοποίηση αυτών των εισόδων. Αλλιώς θα είναι ένα πραγματικό χαράτσι, ένας νέος φόρος που θα ε, επιβαρύνει περαιτέρω τις ε, ευρωπαϊκές μεταφορές. Γι' επαναχρηματοδοτηθουν στι είναι αρκετά επίμαχο αυτό το καταλαβαινα να γινει πραγματικη αξιοποιηση αυτων των εισοδων αλλιω θα ειναι ενα πραγματικο χαρατσι ενα νεο φορο που θα επιβαρυνει περαιτερω τι ευρωπαικε μεταφορε γι αυτο ειναι αρκετα επιμαχο αυτο το θεμα Ευχαριστούμε κύριε Τζανέσκη για ένα λεπτό κύριο Σκράμερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, οι μεταφορέ στην Ευρώπη είναι πολύ φτηνέ, ε, αλλά ε, οι φιλικέ προς το περιβάλλον είναι πανάκριβες. Ε, είναι θελημένο αυτό, αθέμητο ανταγωνισμό που δεν σώζεται με αυτή την οδηγία. Έχουν φορολογικέ ελαφρύνσει και προνόμια τα φορτίγα 60.000 φορές περισσότερο ε, ρηπαίνει ένα φορτηγό από ένα γιοταχή. Δεν είναι αντίστοιχα τα διόδια. Εδώ και δεκαετίες είναι διαφορετική η κατάσταση. Για κάθε χιλιόμετρο, ε, ε, κάθε μηχανή τρένου, ανεξάρτητα από το αν μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα, πρέπει να πληρώνει για κάθε χιλιόμετρο σιδηροδρομικής ράγας στι οδικές μεταφορές αυτό είναι περιορισμένο, αφορά μόνο φορτηγάνο το 3,5 τόνων. Είναι αθέμητος λοιπόν ανταγωνισμός ε, προ όφελο των οδικών μεταφορών που είναι κατά το ε, περιβάλλοντος και ε, κατά του σιδηροδρόμου. Εμείς οι πράσινοι θέλουμε να προστατεύσουμε το κλίμα και να εξασφαλίσουμε στο μέλλον την κινητικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται υγιής ανταγωνισμός και αυτή η Ευρωβινιέτα είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό προς το στόχο αυτό. Ο κύριος Μπάφτον, ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή ε, η διαδικασία ε, τελών ε, στα φορτηγά και στις οδικές μεταφορές είναι κάτι το οποίο τελικά θα επιβαρύνει τον φορολογούμενο και η κυβέρνησή μας προετοιμάζει κάτι για το 2015. Είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός από ξένα φορτηγά που ε, είναι στις διεθνείς μεταφορές και δεν ε, πληρώνουν τίποτα για να χρησιμοποιήσουν τους δικούς μας δρόμους. Ε, ενώ η κυβέρνηση εισπράττει από την αύξηση των καυσίμων. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τέλος μόνο σε ξένα φορτηγά. Ε, αλλά τελικά έχουμε ένα έμεσο φόρο το 2013. Θα πρέπει όμως επειδή είναι φορολογικό το μέτρο να έχει ομοφωνία στο Συμβούλιο. Γίνεται μια προσπάθεια ε, να επιβληθεί έμεση φορολογία χωρίς να το έχει ψηφίσει κανείς σε κανένα δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Ντεβεράκ παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στη στρατηγική της για την Ευρώπη 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο η οικονομία μας να είναι πιο οικολογική και οι μεταφορές πιο σύγχρονες. Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε μεγάλο βαθμό υποστήριξαν αυτό το στόχο συμπεριλαμβανομένων των ε, κρατών μελών και των κοινοβουλίων τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Είναι λοιπόν λυπηρό που από το 2008 και μετά πολλά κράτη-μέλη ε, φέρονται... Ε, να ε, προσπαθούν να ε, μειώνουν την αξία αυτού του προγράμματος και να μπλοκάρουν το πρόγραμμα. Σήμερα, χάρη στην επιμονή του Σαΐντ Ελχατράουι και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και των ε, σχεδόν εισηγητών στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, επιτέλους έχουμε ένα συμβιβασμό ενώπιό μα. Βέβαια, στο κείμενο αυτό είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξο από την αρχική πρόταση, αλλά για πρώτη φορά θα επιτρέψει να ε, εφαρμοστεί στην πράξη αρχή του ρηπαίνων πληρώνει και να εσωτερικευθεί το εξωτερικό κόστο, ε, όπω είναι ο θόρυβο ή ε, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Α μην είναι όμω ένα απλό φόρο η Ευρωβινιέτα να βοηθήσει στη βελτίωση των μεταφορών. Γι' αυτό καλούνται τα κράτη-μέλη να επανεπενδύσουν στον εξυγχρονισμό των μεταφορών τα έσοδα από το τέλο αυτό. Επίση, το Κοινοβούλιο κατάφερε να προωθήσει ε, πολύ τι βελτιώσει στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων διοδίων και με κίνητρα ε, για να χρησιμοποιούμε λιγότερο ρηπαίνοντα βαριά φορτηγά. Και για να είμαστε και σύμφωνοι με τους πολιτικούς μας στόχους, ελπίζω να εγκρίνουμε αυτή τη ε, πρόταση συμβιβασμού σε δεύτερη ανάγνωση και να έχουμε πιο μεγάλη αεφορία στις μεταφορές. Ευχαριστώ, κυρία Ντεβεϊράκ. Για το λόγο κύριο Σπαρνιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτέλους μια ικανοποίηση. Η τιμή του, των διοδίων ε, οδικών μεταφορών με ανώτατο όριο που δίνει οδηγία για την Ευρωβινιέτα θα μπορεί να περιλάβει και το κόστο τη συγχωρήπανση και τη ρήπανση του περιβάλλοντο. Νέα ικανοποίηση είναι ότι με την έκθεση Αρκαντράου και συγχαρητήρια στο ΣαΐΔ για την πυγμή που έδειξε εκφράζουμε, διατρανώνουμε τη θέλησή μας να ε, συμπεριλάβουμε την αρχή ορυπαίνων πληρώνει στη, στο συνυπολογισμό του κόστους των ε, οδικών μεταφορών. Μετά από τριετής διοργανικές διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε σε μια συμβαστική λύση στον τριμερή διάλογο, ώστε πραγματικά να έχουμε μια προστατευτική για το περιβάλλον πολιτική, αλλά ταυτόχρονα και μια αποτελεσματική οικονομική πολιτική σε θέματα ανάπτυξης των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Μία προσοχή όμω, θα πρέπει πραγματικά το, ένα, τμήμα, ένα μεγάλο τμήμα των εσόδων να χρησιμευτούν στι υποδομέ και σε διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, όπω αναφέρεται. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε προ αυτό. Έχω όμω και ε, μία, ε, μία θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου γιατί η αρχή ορυπαίνων πληρώνων δεν ε, γενικεύθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε εκτενώς και παρά την πυγμή που έδειξε ο εισηγητής Σαϊντελ Καντράουι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Επίτροπε, έχασε σε αυτή τη διελκυστίνδα απέναντι στους εθνικισμούς ή τους εθνικούς εγωισμούς, δυστυχώς. Για ένα λεπτό, το λόγο έχει ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την θαυμάσια δουλειά που παρουσίασε σε αυτό το δύσκολο θέμα. Ε, το είπαν αυτό και άλλοι πάρα πολλοί. Ε, τα κράτη-μέλη ε, καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα έσοδά τους ε, για την βελτίωση του περιβάλλοντος. Όταν ε, απευθυνόμεθα στι κυβερνήσει, ε, αυτά τα οποία λέμε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το θέμα δεν είναι να πληρώνουν οι μεταφορεί ε, για τη ρήπανση του περιβάλλοντο χωρί τα χρήματα που συγκεντρώνονται να χρησιμοποιούνται για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτή τα βέβαια τα νέα έσοδα να μην είναι ε, ένα, μια νέα μορφή φόρου όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση να περιοριστούν οι εκπομπές ε, καυσερίων στην Ευρώπη. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα. Για ένα λεπτό κύριος Φαντάλεν. Πρόεδρε, στην απόφαση για την Ευρωβινιέτα ε, πραγματικά είναι ένα ορθό βήμα της Ευρώπης για να εφαρμόσει στις μεταφορές την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Το κόστος για τη χρήση των υποδομών ε, θα πρέπει να συνυπολογίζεται και να καταλογίζεται στο μεταφορέα. Γιατί είναι και η χορύπανση και η ρήπανση με το διοξείδιο του άνθρακα. Ελπίζω να ε, το κάνει η πλειοψηφία των κρατών αυτών και η κυβέρνηση της χώρας μου η ε, κυβέρνηση θα πρέπει να ε, καταλάβει ότι χρειάζεται εφαρμογή και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει προτάσεις έτσι ώστε σταδιακά αυτό το κόστος να εσωτερικευτεί και σε άλλους τρόπους μεταφοράς. Βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του κάθε τομέα. Ας πούμε η εσωτερική ναυσιπλοεία δεν είναι η μόνη ε, ε, που χρησιμοποιεί ε, τις εσωτερικές πλωτές οδούς γιατί είδαμε τώρα με την ξηρασία τι έγινε και πόσο έπεσε η στάθμη των ποταμών γιατί ποτίζουν οι αγρότες. Άρα θα πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη μας. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Το λόγο έχει ο κύριος Δεγκράντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και κάποιες άλλες χώρες συμφωνούν ε, και είναι διστακτικές να δεχθούν το λεγόμενη Ευρωβινιέτα. Κριτική ε, είναι ε, το αποτέλεσμα, αλλά εμείς είμαστε περιφερειακές χώρες και θα πληρώσουμε αυτό το τέλος προς όφελος των κεντροευρωπαϊκών χωρών. Η λογική που είναι πίσω από το τέλος αυτό είναι πολύ αντιφατική. Και κάθε μέρα ε, αποδυναμώνεται η φωνή που το υποστηρίζει. Βέβαια, είναι λογικό να εσωτερικευτεί το εξωτερικό κόστο, αλλά τελικά δεν ευσταθεί αυτό ότι για να, αντιπο... Ε, ε, να αποκριθούμε στην συμφόρηση θα πρέπει να επιβαρύνουν τα βαρέα φορτηγά. Είναι προφανής η διάκριση εδώ στην αρχή του ρηπαίνων πληρώνει. Κατά τα άλλα, η Ευρωβινιέτα θεωρήθηκε στην αρχή ένα είδο χρηματοδότηση των υποδομών, αλλά τελικά μόλι το 15% θα πηγαίνει στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και μάλιστα όχι υποχρεωτικά, αλλά ω απλή σύσταση. Έτσι ώστε ο εκάστοτε υπουργό Οικονομικών θα αποφασίζει τι τον ενδιαφέρει και τι συμφέρει περισσότερο τη χώρα του στο μεγάλο κεφάλαιο των υποδομών. Και το τελικό αποτέλεσμα ε, ε, θα είναι ακόμα περισσότερο άλλη μια φορά άλλο ένα πλήγμα στις οδικές μεταφορές που σήμερα τόσο πλήττονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο ομοίδε σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά δεν χωράει πειραματισμούς που τελικά θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την επισφαλή θέση της οικονομίας μας με επιπλέον κόστος. Τέλος, η επιστική κρίση που σήμερα πλήττει τα ισπανικά προϊόντα ε, έχει ε, προκαλέσει ε, μεγάλη ένταση, άδικη και επιβαρύνει ακριβώς τους ίδιους με την Ευρωβινιέτα και τους μεταφορείς η δική μας αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος Ισπανική τελικά θα καταψηφίσει. Ευχαριστώ κύριε Ντεγκράντε. Στο λόγο έχει για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Δανέλης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Γενική Αρχή που εισάγει η οδηγία στη μεταφορά εμπορευμάτων, η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους, είναι ιδιαίτερη ουσιαστική και συμβολική σημασία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα ευέλικτο πλαίσιο εφαρμογή τη αρχή του ορυπαίνων πληρώνει αλλά και ένα εργαλείο μετριασμού των προβλημάτων συμφόρησης μεγάλων εθνικών αρτηριών. γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να καμφθούν τελικά οι ανησυχίες κάποιες δικαιολογημένες που έχουν εκφραστεί από πολλούς σχετικά με τις ανισομερείς επιπτώσεις της εφαρμογής στην περιφέρεια της ένωσης και στον κλάδο των οδικών μεταφορών. το συμβαστικό κείμενο που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον ε, συνάδελφο αλ σκοπεύει άλλωστε στη σταδιακή εφαρμογή των σχετικών τελών ώστε να συνοδευτεί παράλληλα από μια σταδιακή ανανέωση του ευρωπαϊκού στόλου. αυτό όμως που θα κάμψει τις αντιρρήσεις και θα αποτελέσει προϋπόθεση της αποδοχής αλλά και της αποτελεσματικότητας του πλαισίου της ευρωβινιέτας είναι αφενός η πιστή και διαφανής εφαρμογή της οδηγίας γρήγορα στο σύνολο των χωρών μελών αφετέρου η διοχέτευση του συνόλου των εσόδων ως ανταποδοτικών πόρων στις υποδομές μεταφορών και όχι στο να κλείσουν τις γνωστές μαύρες τρύπες. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δανέλη. Για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πίρκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι το αποτέλεσμα συμβιβασμού, όμως είναι ένας καλός συμβιβασμός. Καλό τον χαρακτηρίζω, διότι ο συμβιβασμό αυτός λαμβάνει υπόψη του και τις δύο πλευρές, τουλάχιστον μέχρι ενός βαθμού. Από τη μια πλευρά λαμβάνει υπόψη του τους μεταφορείς και από την άλλη τους πολίτες οι οποίοι υποφέρουν από την ηχορύπανση και από τα καυσέρια. Τρία τα πλεονεκτήματα της οδηγίας. Πρώτον, τα έσοδα από τα τέλη θα δεσμεύονται για επενδύσεις για τη βελτίωση των μεταφορών. Αυτό από πλευράς οικονομικής είναι πολύ ενδιαφέρον, θα οδηγήσει στη βελτίωση των αρτηριών και ούμονον αυτό θα βελτιωθούν τα έσοδα, ε, θα μειωθεί το κόστος. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι τα κράτη-μέλη αποκτούν τη δυνατότητα το κόστος, ε, τον θόρυβο, ε, τα καυσαέρια, όλα αυτά να τα συμπεριλάβουν στην ε, χρέωση, στα τέλη. Γιατί αρχή, ισχύει αρχή ορυπαίνων πληρώνει, όποιος χρησιμοποιεί καθαρά φορτηγά απλά εξοικονομεί κόστος. Βεβαίως ε, υπάρχουν κατόπιν τούτου κίνητρα έτσι ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση και να ανανεώνεται ο στόλος των αυτοκινήτων. Γνωρίζουμε ότι στις διαπραγματεύσεις δεν κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες, όμως ε, αυτά τα δύο θετικά στοιχεία μπορέσαμε να τα επιβάλλουμε στις διαπραγματεύσεις και κατόπιν τούτου θεωρώ ότι θα οδηγήσουν στο ευκταίο αποτέλεσμα. Εκείνο το οποίο επιθυμώ είναι κατά την εφαρμογή όλων αυτών να μην προκύψει υπερβολική γραφειοκρατία. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο βεβαίως θα πληγεί το τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμπερίληψη ε, των τελών στο ε, εσωτερικό κόστος των διοδίων θα επιτρέψουν την καλύτερη χρήση των υποδομών την εσωτερήκευση του κόστου του εξωτερικού, κάτι που γίνεται και σε άλλους τομείς. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της συμπερίληψης δεσμολογικών φραγμών που θα αυξήσει το κόστος μεταφορών στις περιφερειακές χώρες και άρα θα αυξήσει και το κόστος των μεταφερόμενων προϊόντων. Δεν θα πρέπει η οδηγία να επιτρέπει διακριτική μεταχείριση ανάλογα με την ε, εθνικότητα, την ηθαγένεια του, του μεταφορέα. Το, το αρθρο βέβαια 4K επιτρέπει στα κράτη-μέλη που θεσπίζουν αυτό το σύστημα των διοδίων ή των τελών να προβλέψουν μια αντιστάθμιση. Κάτι τέτοιο όμως θα οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Είναι σημαντικό τα έσοδα που θα προκύψουν από την ε, συλλογή αυτή των διοδίων ή των ε, τελών της χρήσης του εξωτερικού κόστου, να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα έσοδα για την δημιουργία πιο ασφαλών χώρων στάθμευσης. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Ο... Για ένα λεπτό το λόγο ο κύριος Φιράντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο η μεταφορά των εμπορμάτων είναι ε, περισσότερο βιώσιμη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από επενδύσεις ε, στην υποδομή ε, και με την ανανέωση του στόλου, με την ε, χρήση της ροβινιέτας και της αρχής ορυπαίνων πληρώνει. Απλά συγκαλύπτουμε την πραγματικότητα και το γεγονός ότι ορισμένα κράτη αποφελούνται περισσότερο από άλλα. Ας μην ξεχνάμε ότι όσον αφορά στις μεταφορές, εκεί παίζουν μεγάλο ρόλο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλα αυτά χωρίς να προσφέρουμε μια σωστή ε, επαναχρησιμοποίηση των πόρων, την αποδοτικότητα την ε, φιλική διαμόρφωση των μεταφορών. Ε, κατόπιν τούτου όλα αυτά είναι απαραίτητα για αυτή την οδηγία και εμεί θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ μικρό και όσον αφορά την ε, διαλειτουργικότητα θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό και γι' αυτό ίσως η συνδιαλλαγή θα ήταν ο καλύτερος τρόπο για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τι γωνίε οι οποίε εξακολουθούν να εξέχουν. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Μπρόνς. Η προτινόμενη οδηγία ίσως αποτελέσει τη, τη χαριστική βολή στι στις βρετανικές μεταφορές βαρέων οχημάτων που βρίσκονται σε ευθύνους απορία τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα τα... Ε, Αλλοδαπά, αλλοδαπές εταιρείες ελέγχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των βρετανικών μεταφορών. Και Έχουμε όλο και περισσότερου αλλοδαπού μεταφορεί που χρησιμοποιούν αλλοδαπά φορτηγά και ταλίκες που πληρώνουν στι χώρε του ε, πολύ μικρά τέλη αλλά κυριεύουν τι βρετανικέ μεταφορέ. Ε, ε, στη Μεγάλη Βρετανία, εξαιτία του ανταγωνισμού τη αγαπημένη λέξη τη ευρωπαϊκή ορολογία, χάνουν οι Βρετανοί μεταφορεί. Δεν είναι καθόλου θεμητό αυτό ο ανταγωνισμό, γιατί είναι πολύ ψηλότερα τα κόστορα στο κόστο τη Μεγάλη Βρετανία και των τελών και των καυσίμων. Έτσι, παρόλο που τα προτινόμενα τέλη θα εφαρμόζονται σε όλα τα βαρέα οχήματα, το βάρος στη στο βρετανικό κλάδο μεταφορών θα είναι ολέθριο. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιταχθούμε στην έγκριση αυτή τη οδηγίας. Ευχαριστούμε κύριε Μπρός. Ο κύριος Τόρφμαν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι η εσωτερική αγορά είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και αποτελεσματικές μεταφορές. Εγώ όμως ο ίδιος ε, ζω σε μια διαδρομή από την οποία περνάνε 50 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο. Θεωρώ λοιπόν ότι εκτός από το δικαίωμα να έχουμε αποτελεσματικές μεταφορές υπάρχει και το δικαίωμα των ανθρώπων που βρίσκονται κάθοντων όλων αυτών των διαδρομών να προστατεύονται. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση αυτή καλή είναι, μικρό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, αν τελικά χρησιμεύσει στο να πραγματοποιηθούν επενδύσει, έτσι ώστε να βελτιωθεί η προστασία από την ηχορύπανση, να υπάρξουν σύγχρονα φορτηγά, σύγχρονε σιδηροδρομικέ μεταφορές. Αυτό που είναι θετικό είναι ότι στι ορεινέ περιοχέ θα καταβάλλονται αυξημένα τέλη και αυτό είναι πολύ καλό. Ε, αυτό που βρίσκω κάπως προβληματικό είναι ότι εδώ ισχύει η ε, αρχή ε, της ε, προαιρετικότητας, δηλαδή τα κράτη που δεν θέλουν να έχουν την Ευρωβινιέτα δεν δεσμεύονται να την εισαγάγουν. Και αυτό όχι μόνο είναι διακριτική μεταχείρισης βάρος της Ευρώπης, αλλά και ιδιαίτερα προβληματικό για τους ανθρώπους που πλήττονται. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Σκέλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι γενικά η πρόταση αυτή είναι θετική. Είμαστε στην Ευρώπη και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά όσο γίνεται περισσότερο σε όλους τους τομείς και να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα που οδηγούν σε ρήπανση. Και το τέλος, τα βαρέα οχήματα πραγματικά είναι κάτι ε, το οποίο είναι χρήσιμο και λογικό. Κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερα να αναπτύξουμε είναι το εξής. Καλή τεχνολογία αλλά θα πρέπει να βρούμε μια τεχνολογία για τους κινητήρες που να λειτουργούν με λιγότερα καύσιμα, δηλαδή για ε, ε, περισσότερα χιλιόμετρα στο λίτρο. Θα πρέπει να γίνουν πολλά και όχι μόνο για τα βαρέα φορτηγά και για τα υπόλοιπα οχήματα. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει αφαιρθεί, ούτε προωθείται, ούτε γίνεται έρευνα αρκετά εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Και τώρα, ο κύριος Ενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους τίθεται το ερώτημα της φορολόγησης ε, της οδικής μεταφοράς ε, αγαθών και εμπορευμάτων. Η Ευρωβινιέτα είναι καλό για όλους τους Ευρωπαίους. Αλλά έχουμε ακόμα πόρο ε, από το να κάνουμε μεταφορείς να δεχτούν και να πληρώσουν ε, το τμήμα που τους αναλογεί στην κοινωνία. Εγώ ζω σε μια πόλη που περνάνε κάθε χρόνο εκατομμύρια φορτηγά και σας διαβεβαιώ ότι τα δεινά του πληθυσμού λαμβάνονται σπάνια υπόψη. Επίσης κάτι που δεν θέλουμε εδώ να αναφέρουμε τα μεροκάματα του τρόμου ε, των ε, οδηγών. Ε, είναι απαράδεκτη η κατάσταση για την ασφάλεια όλων. Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί είναι στο κάτεργο οι οδηγοί. Θα πρέπει να έχουμε συνδυασμένες μεταφορές με το σιδηρόδρομο μέσω της θάλασσας και των ποταμών με τρόπο ευφυή και σωστό για να μην επιβαρυνθούν ούτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των μεταφορών ε, ούτε οι υποδομές ε, των αυτοκινητοδρόμων ούτε οι ε, μικροί φορολογούμενοι αλλά οι μεγάλοι που δίνουν τις εντολές και τις παραγγελίες. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε τώρα τη συζήτηση ο Επίτροπος κ. Κάλλας έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη, κύριε Πρόεδρε, για τα σχόλιά σας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, η Ευρωβινιέτα δεν είναι ευρωπαϊκός φόρος. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Κατόπιν τούτου, κακό είναι, μάλλον ε, είναι μια οδηγία η οποία περιορίζει και ρυθμίζει τα εθνικά τέλη. Έχουμε 22 ε, κράτη με διαφορετικό σύστημα χρέωσης φορτηγών που χρησιμοποιούν τις οδικές μεταφορές έχουμε βαριά φορτηγά, έχουμε ε, αυτοκίνητα ιδιωτική ε, χρήση. Όσοι ε, χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα μεταφορά πληρώνουν και διαφορετικά τέλη. Δεύτερον που θέλω να πω, παρακαλώ, δεχτείτε το συμβασμό. Γιατί ο συμβασμό είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι φαίνεται. Πίσω από το συμβασμό κρύβονται δύο μάχε. Πρώτον, για την αρχή. Ποιο και γιατί πρέπει να πληρώνει για τη χρήση τη υποδομή. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση ο χρήστης ε, πληρώνει, ε, ισχύει η αρχή ορυπαίνων πληρώνει, θα εξακολουθήσει να ισχύει η σωστή κατεύθυνση. Η δεύτερη μάχη ε, εξακολουθεί να υφίσταται και είναι πολύ πιο οξία. Είναι ένας αγώνας ανάμεσα στις χώρες οι οποίες δέχονται τις, τα βαρέα οχήματα και οι οποίες επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ε, και ε, επιθυμούν να επιμερίζεται το βάρος ε, χρήσης υποδομής ανάμεσα στους φορολογούμενους, στους φορολογούμενους και σε όλους τους χρήστες. Όλοι οι χρήστες, παραλαμβάνομαι, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Και από την άλλη υπάρχει μια ομάδα χωρών κάθετα αντίθετη. Η ομάδα αυτών των χωρών φάνηκε και σήμερα εδώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εγώ απλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στις 15 Οκτωβρίου το Συμβούλιο συμφώνησε ως προς τον πολιτικό συμβασμό. Ε, η μειοψηφία, μάλλον η πλειοψηφία που επιτέχθηκε ήταν οριακή και ο αγώνας συνεχίζεται. Ο εισηγητής έκανε μια θαυμάσια δουλειά, αγωνίστηκε για να επιτύχει έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό και να καταθέσει μια καλή πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν σας κάνω έκκληση ειλικρινά. Παρακαλώ στηρίξτε αυτό το συμβιβασμό ε, πολλές ε, λεπτομέρειες ίσως να μην είναι ικανοποιητικές ε, για διάφορους εμπλεκόμενους και άλλους είναι όμως ένα μεγάλο βήμα το θέμα υπάρχει, χρονίζει εδώ και χρόνια και τώρα να, ειδού η ευκαιρία για να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, το λόγο έχει η κυρία Γκέρι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πολύ αξιόλογη συζήτηση. Αναφέρθηκαν ε, πολλά επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα και όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ έχουμε έναν πραγματικό συμβασμό παρά τις ε, δυσκολίες ε, που προέκυψαν. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι είναι μια αμυγής ε, ευρωπαϊκή επιτυχία, όπως είπε και ο κύριος Λάιχτφριτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για την Ουγγρική Προεδρία, όπως και σε κάθε συμβασμό και αυτό είναι το αποτέλεσμα ισορροπιών. Αναζητήσαμε την ισορροπία ανάμεσα σε επιχειρήματα υπέρ του περιβάλλοντος και ανάμεσα σε άλλα υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης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 το περιβάλλον είναι σημαντικό ε, για το Συμβούλιο. Γιατί αν δεν ήταν, δεν θα είχαμε τελικά και αυτήν την οδηγία. Ε, θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μια φορά αυτή την ισορροπία ανάμεσα στις χώρες του κέντρου και αυτές της ε, περιφέρειας. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση για το πώς μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε μια λύση που θα ωφελεί και τις χώρες περιφέρειας να μην αισθάνονται αυτές παραγωνισμένες. Μεγάλη συζήτηση για το πώς θα βρούμε μια ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Ε, ίσως Αυτά όλα να είναι σταγόνα το ωκεανό, αλλά εγώ παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση εσωτερήκευσης του εξωτερικού κόστους ε, και ε, προς την κατεύθυνση της ε, διοχέτευσης ε, κονδυλίων προς τις μεταφορές. Εφόσον είναι συμβασμός, προφανώς και δεν είναι τέλειος και γι' αυτό λοιπόν ελπίζω κατά τα επόμενα έτη να μας προσφερθεί η ευκαιρία να βελτιώσουμε αυτό το συμβιβασμό. Όσον αφορά στα θέματα, επί της ουσίας δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει το θέμα των εσόδων. Ε, η χρήση των εσόδων που θα προκύψουν από τη συγκέντρωση των τελών. Στη συμφωνία ε, προβλέπεται λεπτομερώς μια σύσταση για τα κράτη-μέλη για το πώς καλούνται να χρησιμοποιήσουν ε, τα έσοδα αυτά τουλάχιστον 15% αυτών των εισόδων, όπως είπε και η κυρία Μάιστερ, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός ε, πολύ καλού συμβιβασμού και όπως ε, αναφέρθηκε ήδη, ίσως να είναι μόνο το πρώτο βήμα, αλλά τουλάχιστον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το δεύτερο θέμα, ετέθηκε αυτό από τον κύριο Στέρξ, ε, σχετικά με το κόστος ε, συμφόρησης. Η συμφωνία καλύπτει και αυτό το πρόβλημα, διότι δίνει τη δυνατότητα στα κρατημέλη να επιβάλλουν τέλη και να ε, διαφοροποιούν ε, ως προς το ύψος ε, των τελών ανάλογα με τον τόπο και το χρόνο. Έτσι λοιπόν τα κρατημέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν υψηλότερα τέλη κατά τις περιόδους συμφόρησης και τις ώρες εχμής. Ε, είναι λοιπόν μια εναλλακτική λύση, ένας ε, τρόπος για να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση, οποτεδήποτε προκύπτει αυτή. Αν λαμβάνεται ε, μόνο η ρήπανση στο εξωτερικό κόστος, ε, ακόμα και έτσι οι μηχανισμοί διαφοροποίησης μπορούν να συμβάλλουν στο να περιορίζονται οι ε, συμφορήσεις στις ευρωπαϊκές αρτηρίες. Το τελικό ερώτημα ετέθη από τον κύριο Λίχτενμπεργκ σχετικά με το εξωτερικό κόστος το Συμβούλιο στις 14 ε, ε, Δεκεμβρίου στην πρώτη ανάγνωση κατέληξε ως προς τη θέση του και κατόπιν μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου προβλέψαμε μία διάταξη στην οδηγία για να εκπέμψουμε πολιτικό μήνυμα προς τους ε, πολίτες. Έτσι λοιπόν συμπεριλάβαμε στην οδηγία μία διάτοξη σύμφωνα με την οποία ε, στις ορεινές περιοχές ε, μπορεί να επιβάλλεται ένα επιπρόσθετο κόστος γιατί οι κατηγορίες αυτοκίνητων ε, υπαριθμών 3 ρηπαίνουν περισσότερο από άλλες κατηγορίες της κατηγορίας 1 και 2. Εξάλλου, για να ενισχύσουμε την ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων. Ε, προβλέπουμε κίνητρα για αυτοκίνητα κατηγορίες 5 και 6 που ρηπαίνουν λιγότερο. Αυτός είναι ένας στόχος που ε, θα επιδιώξει η οδηγία. Αγαπητά μέλη, ε, κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση κατέστησε σαφές ότι η οδηγία για την Ευρωβινιέτα είναι ένα θετικό και σημαντικό βήμα για τον τομέα των μεταφορών. Η πρόταση για τα βαρέα οχήματα είναι και αυτή πολύ σημαντική, αλλά είναι και συμβολική. Γιατί είναι η πρώτη φορά, και το είπατε και εσείς αυτό, είναι λοιπόν η πρώτη φορά που τίθεται σε εφαρμογή η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Εμείς λοιπόν επιθυμούμε να εσωτερικεύσουμε το εξωτερικό κόστος σε όλα ε, σε όλες τις μεταφορές στο μέλλον. Η Ουγγρική Προεδρία είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για το ότι ε, κατέληξε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι πεπισμένη ότι τα μέτρα ε, που θα προτείνει το Κοινοβούλιο θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα και σε φιλικότερες μεταφορές προς το περιβάλλον και κατόπιν τούτου οι πολίτες ε, θα είναι οι τελικοί ωφελημένοι από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ και για να τελειώσει ε, τώρα έχει το λόγο ο εισηγητής ο κ. Αλχαντραό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξη ε, και τα σχόλια και εκείνων που διαφωνούν. Είναι πολύ σημαντικός ο τομέας των μεταφορών για την οικονομία μας, αλλά προκαλεί και κάποιο κόστος, όχι μόνο για την υποδομή. Έχουμε σωματίδια στην ατμόσφαιρα, ε, συμφόρηση, θόρυβο, ηχορύπανση. Τώρα επιτέλους έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη ε, να χρεώνουν ένα μερίδιο του κόστους στον ρηπαίνοντα για να έχουν και μέσα και έσοδα ε, επανεπένδυσης ε, ανταποδοτικά στο σύστημα των μεταφορών για να ε, μειωθεί το κόστος και να βελτιωθεί η λειτουργία της κοινωνίας, η αποτελεσματικότητα του κλάδου και να συνεισφέρουμε και λίγο για ε, καλύτερους ε, τρόπους ε, και ίσους όρους παιχνιδιού των διαφορών μέσων μεταφορών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτή την πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο φιλοδοξεί το 2020 να είναι υποχρεωτική η Ευρωβινιέτα και αυτό υπόσχεται πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το μέλλον. Πάντως βλέπω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, ε, έχουμε αρκετή στήριξη ε, από την Ολομέλεια για να δείξουμε ότι η Ευρώπη παίρνει αποφάσεις προς όφελος των πολιτών της. Ελπίζω κάποιες χώρες τώρα να εφαρμόσουν αυτή τη δυνατότητα ε, που ανοίγεται και να έχουν καλά αποτελέσματα για να συμπαρασύρουν και άλλες χώρες στην κατεύθυνση αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και ευρύτερη υποστήριξη για να προχωρήσουμε και αποδοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τώρα έχει πολλή δουλειά με αυτή την οδηγία για να κάνει έρευνα τις άλλες ε, παραμέτρους ε, του εξωτερικού κόστους, αν μπορούμε τα επόμενα χρόνια να τα συμπεριλάβουμε, αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος. Ε, σήμερα έχει γίνει ένα πρώτο βήμα και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χαντράουι. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ακολουθούν οι ψηφοφορίες.